Uh, dear colleagues, good afternoon. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Continued meeting of the Committee Καλώς ορίσατε στην απογευματινή συνεδρίαση της Επιτροπής ε, Νομικών Υποθέσεων. Συνεχίζουμε με το σημείο 11. Εργαστήριο για την Οδηγία για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, ενίσχυση της θέσης των εκδοτών και των δημιουργών και ερμηνευτών εκτελεστών. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους σε αυτό το εργαστήριο, το οποίο διοργανώνει το Τμήμα Πολιτικής ΣΥ θα αναφερθούμε στην οδηγία για τα πνευματικά δικαιώματα που, που συζητούνται αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή μας και πιο συγκεκριμένα σε δύο σημεία της πρότασης αυτής. Πρώτον, στην προτινόμενη δημιουργία ενός νέου δικαιώματος για εκδότες τύπου και δεύτερον στις πτυχές που σχετίζονται με τη δίκαιη αμοιβή ε, για συμβόλαια με ε, δημιουργούς και εκδότες. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε πολλές διαφορετικές απόψεις διαφόρων ακαδημαϊκών ε, του καθηγητή Λάνελ Μπέντλι από το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, τον ε, καθηγητή Μάρτιν Κρίτσμερ από το Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης, τον καθηγητή Τόμας Χάπνερ από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μπελβάου και τον καθηγητή Κρίστοφ Κάρεν, Καρόν, συγγνώμη, από το Παρεπιστήμιο Παρί Εστ Οι προσκεκλημένοι μας θα κάνουν τις παρουσιάσεις τους ε, βάσει του έργου τους και θα απαντήσουν και ερωτήσεις, σε ερωτήσεις των μελών. Σκοπός αυτού του εργαστηρίου είναι να γίνει μια σε βάθος συζήτηση με ακαδημαϊκούς γι' αυτό τα πολύ τεχνικά ζητήματα. Χωρίς άλλη καθυστέρηση θα ήθελα να καλωσορίσω τους ομιλητές μας και δίνω το λόγο στους καθηγητές Λάινελ Μπέντλε και Μαρτίν Κρέτσμερ να μας παρουσιάσουν τις μελέτες τους. Δέκα λεπτά για τον καθένα σας ή 20 λεπτά όλοι μαζί και οι δύο μαζί. Ε, από εσάς εξαρτάται αν θα μοιραστείτε αυτά τα 20 ε, λεπτή χρονοθυρίδα. Κύριε Κρέτσμερ, έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ. Είμαι ο Λάινελ Μπέντλε. Θα παρουσιάσω ε, αρχικά τα δικαιώματα των εκδοτών τύπου. Θα σας περιγράψω κάποιες από τις επικρίσεις που έχουν γίνει για τα δικαιώματα αυτά και στη συνέχεια ο καθηγητής Κρέτσμπερ θα εξηγήσει κάποιο από το εμπειρικό έργο που έχουμε επιτελέσει στο πλαίσιο αυτής της μελέτης αφορά το πώς έχουν εφαρμοστεί οι πρόδρομοι αυτών των δικαιωμάτων στην Γερμανία και στην Ισπανία. Μετά από αυτό θα αφιερώσω λίγο χρόνο στην παρουσίαση των διατάξεων για τις αποζημιώσεις των ε, δημιουργών. Δηλαδή θα αφιερώσουμε 15 λεπτά για τα δικαιώματα των ε, εκδοτών τύπου και 5 λεπτά για τις αποζημιώσεις των δημιουργών. Αλλά ευχαριστώ φυσικά να απαντήσουμε σε ερωτήσεις στη συνέχεια. Δυσκολεύομαι να διαβάσω και το δικό μου PowerPoint φοβάμαι, αγαπητοί κύριοι. Μια γρήγορη υπενθύμηση για το πού βρισκόμαστε. Η Κομισιόν υπέβαλε μια πρόταση για τα διανοητικά δικαιώματα στην ενιαία αγορά το Σεπτέμβριο του 2016. Η πρόταση εξετάστηκε από διάφορε επιτροπέ. Ήρθε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μια πρώτη ανάγνωση και τώρα μελετάτε και έχουν συνταχθεί και σχετικές εκθέσεις ε, από ε, τις Επιτροπές ΕΜΚΟ ή και πρέπει να περάσει και από αυτήν εδώ την Επιτροπή. Αυτό έχει προγραμματιστεί κάποια στιγμή τον Ιανουάριο. Ταυτόχρονα εξετάζεται με την κανονική διαδικασία ε, στο Συμβούλιο και αυτή τη στιγμή έχουμε και κάποιε διαφορετικέ διατάξει τη προτάσει, τι συμβαστικέ προτάσει τη Εστονική Προεδρία που δημοσιεύθηκε τέλη Αυγούστου. Ας ξεκινήσουμε με τα δικαιώματα των εκδοτών τύπου. Μα ζητήθηκε από μια επιτροπή να κάνουμε μια αναθεώρηση των ακαδημαϊκών επικρίσεων που έγιναν επί αυτών των δικαιωμάτων αρκετά ευρύε επικρίσει. Μα ζητήθηκε επίση να δώσουμε κάποια εμπειρικά αποδεικτικά στοιχεία για την τρέχουσα κατάσταση στη Γερμανία και την Ισπανία. Το δικαίωμα θεσπίζεται με το άρθρο 11 της πρότασης, όπου η Κομισιόν εξηγεί ότι υπάρχουν δύο στόχοι. Ότι επιτελεί δύο στόχους. Πρώτον, διασφάλιση βιώσιμου τύπου, κάτι που όλοι στον ελεύθερο κόσμο θεωρούν αξιοθαύμαστο στόχο. Ε, δεύτερον, διευκολύνει τους εκδότες να συνάπτουν άδειες και να εφαρμόζουν δικαιώματα. Η Κομισιόν δίνει ένα παράδειγμα γερμανικό, όπου ένας εκδότης τύπου συγκέντρωσε τις άδειες ε, και τα αποκλειστικά δικαιώματα 20.000 ε, εκδοτών ε, για να μπορέσει να προβεί σε δράση στη Γερμανία. Η απάντηση της Κομισιόν στα εν λόγω προβλήματα ήταν τα δικαιώματα ε, εκδοτών τύπου που ορίζονται στο άρθρο 2 με πολύ γενικό λόγο τρόπο. Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιες διαφωνίες όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή που καλύπτεται από αυτό το δικαίωμα των εκδοτών τύπου, οι οποίοι θα απολαύουν του δικαιώματο αναπαραγωγή ενό έργου και διάθεση του στο κοινό. Ωστόσο, το δικαίωμα αυτό περιορίζεται εντό τη πρόταση σε ψηφιακέ εφαρμογέ. Θα έχει διάρκεια 20 ετή και θα υπόκειται στι εξαιρέσει στις οποίες μπορεί να υπόκειται τα πνευματικά δικαιώματα και το copyright και η οδηγία για το, και το άρθρο 5 της οδηγίας για το copyright ε, δίνει το περιθώριο στα κράτη-μέλη για συγκεκριμένε εξαιρέσει που θα εφαρμόζονται ε, στο δικαίωμα διανοητική ιδιοκτησία και τα σχετικά δικαιώματα και τα συναφή δικαιώματα. Οι ακαδηματικές επικρίσει λαμβάνουν δύο μορφέ. Πρώτα απ' όλα, ένα προβληματισμό ε, όσον αφορά το τι έχει σχεδιαστεί να επιτύχει το δικαίωμα. Και αυτό συνοψίζεται σε δύο ερωτήσει. Πρόκειται για δικαιώματα που αλλάζουν την ουσία των όσων έχουν ήδη στη διάθεσή τους οι ε, εκδότες τύπου ή ο σκοπός είναι να αποκτηθεί ένα δικαίωμα σαν αυτό των ε, δημιουργών. Δηλαδή από τη μία απόψη, εάν η ουσία, επί της ουσίας το δικαίωμα δεν διαφέρει ιδιαίτερα, τότε δυσκολεύεται κανείς να καταλάβει τι θα επιτύχει ε, αν θα βελτιώσει τη θέση των εκδοτών τύπου. Οπότε πρώτος στόχος της ε, Κομισιόν ε, όντας ε, ο βιώσιμος τύπος. Το ερώτημα είναι ότι αν δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά επί της ουσίας πώς θα επιτευχθεί αυτό. Εντάξει, επί των τύπων δεν είναι διαφορετικό. Λέει απλά ότι οι εκδότε τύπου θα έχουν διάφορα δικαιώματα που έχουν αναγνωριστεί στο πλαίσιο τη οδηγία για την κοινωνία πληροφοριών. Και ότι θα, σε αυτά τα δικαιώματα θα εφαρμόζονται κάποιε εξαιρέσει. Οπότε ανακύπτει το ερώτημα, τα δικαιώματα αυτά είναι, έχουν διαφορετικό πεδίο εφαρμογή και πολλοί εμπειροί εδώ, εμπειρογνώμονες εδώ θεωρούν ότι υπάρχει κίνδυνος κάποιοι θα έλεγαν όφελος ε, διότι υπάρχει διαφορά στην ουσία στο πεδίο εφαρμογή. Ουσιαστικά, σε περίπτωση παραβίασης του δικαιώματος δημιουργού, παραβιάζει ε, πραγματικά, η παραβίαση μόνο ε, όταν η παραβίαση αφορά τη γνησιότητα του έργου. Δηλαδή, παραβιάζει κανεί τα διανοητικά δικαιώματα ε, σε ένα δημοσιογραφικό άρθρο αν πάρει ένα κομμάτι το οποίο είναι το ε, original, που είναι το αρχικό. Αλλά το δικαίωμα που δίνεται εδώ είναι ένα συγγενές δικαίωμα. Δεν σχετίζεται με αυτή την απέτηση γνησιότητας ε, αρχικής έκδοσης. Οπότε αναρωτιέται κανείς κατά πόσο αυτό θα επεκταθεί σε μικρότερα τεμάχια υλικού ε, όπου θα εντάσσεται στα παραδοσιακά δικαιώματα δημιουργού. Τι γίνεται δηλαδή με αυτό που ονομάζεται αποσπάσματα, snippets ή και συνδέσεις, ε, τα links. Διότι και τα links είναι σύντομα αποσπάσματα ουσιαστικά. Είναι πολύ εύκολο να κάνει κανείς ένα link προς μια πρόταση, ένα τίτλο ενός δημοσιεύματος και αν αυτό θεωρηθεί snippet, αν θεωρηθεί απόσπασμα, τότε και τα links αυτά, οι συνδέσεις θεωρούνται και αυτές μικρά αποσπάσματα. Εάν συμβαίνει αυτό και το εάν αυτό είναι μεγάλο, δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι κατά πόσο υπάρχει πρόθεση να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογή ε, τη προστασία και σε αυτό το δικαίωμα, αυτό θα δημιουργήσει σημαντικέ δυσκολίε. Αφενό, δεν είναι απόλυτα σαφέ ποιο κριτήριο θα χρησιμοποιείται για να πιστοποιηθεί η παραβίαση. Δεύτερον, θα υπάρξουν συνέπειε όσον αφορά την ελευθερία έκφραση. Αν απαγορεύσουμε στου ανθρώπου να χρησιμοποιούν πολύ μικρά κομμάτια κάποιου έργου ειδικότερα αν το έργο αυτό είναι ιδιαίτερα μεγάλο Είναι σοβαρά λοιπόν τα προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν δομικά δηλαδή. Δεύτερον, αν υπησέρχεται αλλαγή, μεταβολή τη ουσία, έχουμε τι εμπειρίε από την Ισπανία και τη Γερμανία που θα εξηγήσω ο Μάρτιν σε λίγο. Όπου λέμε ότι ακόμη και αν επεκτείνουμε τα διανατικά δικαιώματα, οι επιπτώσει δεν θα είναι και μεγάλε, αν έχει αλλάξει κάποιο ελαφρώ το κείμενο. Το θέμα είναι τώρα εδώ κατά πόσο η πρόταση αυτή προτίθεται να δώσει ένα δικαίωμα ίσο με αυτό των συγγραφέων και στους εκδότες όπου εκεί λοιπόν η πρόταση είναι να δοθεί ένα δικαίωμα αλλά το αποτέλεσμα δεν θα αφορά επέκταση του περιεχομένου αυτού του δικαιώματος. Αυτός είναι ο στόχος. Η ακαδημαϊκή επίκριση επί αυτής της ιδέας είναι ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί πολύ πιο εύκολα χωρίς να δοθεί κανένα δικαίωμα στους εκδότες. Υπάρχει ένας λιγότερο διεισδυτικός τρόπος ε, παρέμβασης θα μπορούσε να υπάρχει κάποιο τεκμήριο, τεκμήριο ε, ιδιοκτησίας, αντιπροσώπευσης που θα δίνει το δικαίωμα στους ε, εκδότες να ε, κατέχουν τα δικαιώματα που τους ανήκουν στα έργα τα οποία δημοσιεύονται στα δικά τους δημοσιεύματα τύπου. Αυτή είναι η ακαδημαϊκή επίκριση. Αυτό έχει συζητηθεί σε διάφορες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με διάφορους τρόπους. Κάποιες επιτροπές ε, εκδηλώνουν επιφυλάξεις για την πρόταση και κάποιες άλλες θέλουν την επεκτείνουν. Και επίσης ε, παρουσιάζουμε ίδιες ε, διαφορέ απόψεων και εντός της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου, όπου υπάρχουν δύο επιλογές. Η πρώτη είναι εξάλληψη της δυνατότητας ελέγχου των αποσπασμάτων, πραγματική, και η άλλη επιλογή είναι να υπάρχει το τεκμήριο ιδιοκτησία, το οποίο είναι και αυτό που προτείνεται στο σχέδιο έκθεση τη Γιούρη. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Μάρτιν για να σα εξηγήσει τι συνέβη στη Γερμανία και στην Ισπανία. Uh, Γεια σας, ονομάζομαι Μάρτιν. Germany and in Spain. The operation and the effect of the existing press publisher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 και για τα VG Media φτάσαμε στην κατάσταση που δεν ήταν δωρεάν η αδειοδότηση, ήταν υποχρεωτική και άρα κανείς δεν μπορούσε να εξαιρεθεί. Να δούμε τώρα τι έγινε στην ε, Ισπανία. The situation is, is, uh, Είναι δύσκολο εδώ να δούμε ακριβώς πώς έγιναν τα πράγματα. Δεν πρόκειται για νέο δικαίωμα. Έχουμε τροποποίηση στις εξαιρέσεις των συλλογικών αδειοδοτήσεων. Δεν πρόκειται μόνο για νέο δικαίωμα. Αλλά πρόκειται για έναν τρόπο το πώς θα πληρώσει κανείς για να χρησιμοποιήσει αυτά τα μη σημαντικά αποσπάσματα ο σκοπός ήταν ενημερωτικός και υπάρχει εδώ το στοιχείο της υποχρεωτικότητας επομένως που απουσιάζει όσον αφορά τη γερμανική ρύθμιση στην ε, ρύθμιση μας στην Ισπανία μέσα στα τα δυόμιση χρόνια είπαμε ότι δεν είχαμε κάποιες αντιδοτήσεις και φέτος ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις 5 ευρώ για κάθε χρήστη. Και είπαμε ότι έτσι αυτοί που μαζεύουν τα νέα, αυτές οι πύλες, θα πρέπει να πληρώσουν ανάλογα με το πόσοι χρησιμοποιούν το website. Αυτό σημαίνει ψηλό κόστος. Και 2,4 εκατομμύρια ήταν το κόστος που να καταβληθεί. So details about the licensing Αυτά όσον αφορά την κατάσταση για τις αδειοδοτήσεις και τώρα έχουμε μια αδειοδότηση στην Ισπανία για κάποια joint venture μεταξύ δύο ομίλων για την παροχή κάποιων υπηρεσιών προς κινητά τηλέφωνα. Ουσιαστικά έγινε η αδειοδότηση μεταξύ δύο εταιριών του ιδίου μήλου. Τώρα. Ένα άλλο στοιχείο. Το αφορούσε τους εκδότες. Αυτούς τους πάντων μας μίλησαν, γιατί δεν μιλήσαμε σε όλους. Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα από την επαφή μαζί τους. Τώρα εδώ βλέπουμε ότι η αγορά είναι πάρα πολύ δυναμική και οπότε έχουμε σημαντικές αλλαγές όσον αφορά τη μελέτη επιπτώσεων και υπάρχει πτώση όσον αφορά τις ε, συνδρομές και επομένως υπάρχει και μείωση όσον αφορά ε, τις ε, διαφημίσεις στις πλατφόρμες. Πάντως ε, καινούργια μοντέλα αναδύονται. Όπως ο Guardian υπάρχουν κάποιες προσωπικές υπηρεσίες όπως το Alexa του, της Amazon περίπλοκο το τοπίο κάποιοι εκδοτικοί εκεί τα πάνε καλά, κάποιοι όχι. Ας πούμε αυτός ο όμιλο είπε στην τελευταία ετησία έκθεση ότι έχει τζίρο 3,3 δις. Αύξηση 10,7% για το 16. Αυτά για τον Όμιλο Σπρίγκερ. Αυτά μας είπαν οι εκδότες ότι είναι πάρα πολύ ρευστή η κατάσταση. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να μεταβληθεί. Επίσης άλλο συμπέρασμα είναι ότι αυτά είναι στα όνειρα του ωκεανού. Πάμε στα 20 δις ετησίως, 10.000 ετησίως, άμα δείτε σε σχέση με το 3,3 τζίρο, τζίρο ετήσιο, θα καταλάβετε ότι είναι δεκάρες Άλλο συμπέρασμα. Να δούμε τι άλλο έχουμε. Έχουμε κάτι που καθορίζει την εκτοκινή του Ιντερνετ. Δηλαδή θα πρέπει να ξέρει κανείς πού το πάει ένα σύνδεσμος για να μπορέσει να ε, τον αξιοποιήσει, για να λειτουργήσει. Και αν ε, έχουμε μόνο πάρα πολύ μικρά κείμενα που είναι αποδεκτά, και βλέπουμε τι αποφάσισε το Δικαστήριο Σημάτων βλέπετε ότι πολλές φορές η διεύθυνση του Ιντερνετ ή μάλλον ο σύνδεσμος έχει πιο πολλές λέξεις από όσο το κείμενο στο οποίο οδηγεί. Και από ό,τι μας είπαν οι εκδότες ότι αυτά όλα είναι απειλή για την καινοτομία. Το σύστημα στην Ισπανία είπαμε είναι υποχρεωτικό και έχουμε επομένω αυτές τις πύλες και εκεί υπάρχουν κάποιοι στου οποίους οδηγούν οι σύνδεσμοι. Και αν κάποιο είναι νεοφύης επιχείρηση στην Ισπανική αγορά και θέλει έναν τέτοιο, τέτοιο σύνδεσμο δεν μπορεί να το κάνει εάν δεν πληρώσει. Και το θέμα τι γίνεται με τον ανταγωνισμό για το Google και το Facebook στην Ευρώπη. Όχι πώς το κάνουμε με την αδειοδότηση, είναι ακόμα πιο δύσκολο να μπορούμε να φτιάξουμε τις δικές μας πλατφόρμες που να είναι ανταγωνιστικές. Τέλος, οι μεγάλοι παίκτες ήδη κάνουν deal. Ας πούμε στην Ισπανία η Ελπαΐς έκανε με το Facebook μια συμφωνία όσον αφορά τη χρήση του περιεχομένου και πολλά χρήματα αλλάξανε χέρια. Συμπερασματικά βλέπετε εδώ το δείγμα Επομένως είναι άσχετο με το copyright αυτή η μεγάλη στραβή που έγινε και ε, έχουμε μέσα αυτά τα έσοδα τα οποία δεν είναι αποτέλεσμα ε, του copyright. Μεγάλη αλλαγή σε αυτή την τεχνολογία. Δεύτερον, από την ισπανική και γερμανική εμπειρία δεν υπάρχει σαφής ωφέλεια για την οικονομία ή την κοινωνία με τη θέσπιση των νέων δικαιωμάτων. Δεν υπάρχουν αποδείξεις για ωφέλεια σαφή. Τρίτον, εκδότες και δημοσιογράφοι δεν θέλουν το σύστημα αυτό, αυτά τα δικαιώματα. Επομένως, το λόμπι κυριαρχείται από κάποιες, κάποιους λίγους εκδότες. Όχι, όχι οι δημοσιογράφοι που ασχολούνται με το ίντερνετ. Για να μην στριμωχτεί το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μειονεκτική θέση. Δηλαδή, το σύστημα θα πρέπει να το ξαναδούμε αφού είχε, αν έχει αποδώσει σε Ισπανία και Γερμανία. Ένα λεπτάκι για τις ε, συμβατικές διατάξεις. Υπάρχουν τρία είδη. Πρώτον, μηχανισμός διαφάνειας. Δεύτερον, μηχανισμός προσαρμογής της σύμβασης. Και τρίτον, ε, υποχρέωση κρατών μελών να υπάρχουν εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών. Η βασική κριτική μας είναι ότι ε, δεν είναι αρκετά φιλόδοξη αυτή η πρόταση, δεδομένου ότι πολλά έχουν προχωρήσει περαιτέρω. Θα μπορούσε λοιπόν κανείς να σκεφτεί ότι σε εύλογο χρονικό διάστημα θα ήταν σωστό να προταθούν πιο φιλόδοξα μέτρα από αυτά που συζητούμε αυτή τη στιγμή όλα αυτά, στη βάση της περιπλοκότητας της νομοθεσίας διαφόρων κρατών μελών που διέπουν, για παράδειγμα, την, την, την αμοιβή, τη δίκαιη αμοιβή, ε, δεν θα ήταν σωστό να υπάρχει αυτή τη στιγμή μια τέτοια διάταξη χωρίς να έχει υπάρξει διαβούλευση ε, και εκτίμηση του πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί στην πράξη κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Τόμας Χέπνερ, τον καθηγητή, που θα μας παρουσιάσει τη δική του οπτική για το ζήτημα που συζητούμε σήμερα. Δέκα λεπτά έχετε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Πρωτού ε, ξεκινήσω, πρέπει να σας πω ότι δεν είμαι τελείως αμερόληπτος, γιατί στο παρελθόν εκπροσωπούσα εκδότες, όχι όμως το ζήτημα της ε, πνευματικής ε, ιδιοκτησίας. Γιατί το είπα και γιατί ε, με έχετε προσκαλέσει. Νομίζω το γεγονός ε, αυτό οφείλεται στο ότι και οι εκδότες δεν είναι αμερόληπτοι στο θέμα αυτό. Αυτό όμως δεν έχει γίνει ευρύτερα γνωστό. Γιατί, διότι δημόσια ε, είχαν εκφράσει την κριτική του το 2006 στο δικαίωμα των εκδοτών. Μάλιστα στο Ηνωμένο Βασίλειο ξεκίνησαν μια εξαρτία για να, για να σταματήσει αυτή παρα... η πρόταση και αντιτίθενται σε αυτή την πρόταση ε, έκτοτε. Στην πραγματικότητα λοιπόν ε, η ίδια η, η κριτική τους είναι αυτή που έχει επιστρέψει και στον εαυτό τους δηλαδή. Το 2015 αποδείχθηκε ότι η Google, ο μεγαλύτερος ε, πολέμιος αυτής της πρότασης, έχει ε, χρηματοδοτήσει 300 πανεπιστημιακούς ε, για να εκπονήσουν μελέτες υπέρ της. Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι απόψεις αυτών των ε, εκδοτών ε, βασίζονται σε μια εσφαλμένη παραδοχή. Ισχυρίζονται λοιπόν ότι το δικαίωμα των εκδοτών ταυτίζεται με τα πνευματικά δικαιώματα των εκδοτών. Και αυτός είναι ο λόγος που το δικαίωμα του εκδότη δεν θα βοηθήσει κανέναν κατά τη γνώμη τους. Αυτό ισχυρίζονται. Επίσης, αυτοί άλλωστε χρησιμοποίησαν πρώτη φορά την, ε, την, ε, την ιδιότητα του, του, του εκδότη Φυσικά δεν λέω ότι οι πανεπιστημιακοί δεν μπορούν κάποια στιγμή να αλλάξουν και άποψη σε σχέση με παλιότερε δημοσιεύσει του και να είναι ανοιχτοί σε αντεπιχειρήματα, αλλά διαβάζοντα τη μελέτη αυτή, νομίζω ότι αυτή δεν ήταν η προσέγγιση που υιοθετήθηκε από του συντάκτε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για το πόσο μονόπλευρη είναι η μελέτη. Δεν υπάρχει ούτε μία ανάλυση των οικονομικών στοιχείων που σχετίζονται με την ε, ε, οικονομική σχέση ανάμεσα στους εκδότες ειδήσεων και τους aggregators. Μάλιστα ε, υπάρχει ο ισχυρισμός ότι οι εκδότες ειδήσεων ε, ωφελούνται κιόλα από το, την ύπαρξη των aggregator. Δεν υπάρχει όμως καμία εμπειρική απόδειξη ούτε στοιχείο για αυτό που ε, εκείνοι ονομάζουν εμπειρικό τμήμα. Αυτό ε, αυτό το εμπορικό τμήμα βασίζεται απλά σε 8 συνεντεύξεις. Ενώ υπάρχουν 200 εταιρείε που εκπροσωπούνται από την VG Media. Χωρίς όμως να υπάρχει κανείς ε, παρά μόνο αρχισυντάκτες. Αρχισυντάκτες όμως είναι δημοσιογράφοι οι οποίοι υποστηρίζουν αυτό το, το, το δικαίωμα ακριβώς γιατί ε, ωφελούνται έμεσα από το δικαίωμα αυτό. Ταυτόχρονα παρατηρώ ότι στη μελέτη, στη μελέτη ε, αναφέρονται περισσότεροι CEO, διευθύνοντες σύμβουλοι, aggregators παρά εκδότες. Η γερμανική ε, εταιρεία συλλογής η Φάουγκε Μίντια που ισχυρίζεται ότι είναι πεπισμένη ότι αυτό θα λειτουργήσει το δικαίωμα δεν, δείχνει, δεν δίνει κανένα στοιχείο για να στηρίξει αυτόν τον ισχυρισμό της. Επίσης δεν αποκαλύπτεται ότι η κριτική της μελέτης είναι η κριτική που έχουν χρησιμοποιήσει οι ίδιοι συντάκτες και ότι η πανεπιστημιακή αυτή άλλωστε ήταν και μεταξύ εκείνων που πρώτη-πρώτη του 2016 είχαν ε, εκθέσει την ε, διαφωνία τους ε, εξισώνοντας τα, τα δικαιώματα των, εκδοτών και, των, και της πνευματικής ιδιοκτησίας. Από εκεί και πέρα. Έχει αναφερθεί το αν θα πρέπει να καλύπτονται τα αποκόμματα τύπου ή όχι. Κατά τη γνώμη μου είναι σαφές ότι πρέπει να καλύπτονται, διότι αν δείτε τα οικονομικά στοιχεία, εκεί είναι όλο το ζουμί. Το ζουμί είναι ότι σήμερα δεν μπορείς να εκπληρώσεις το κριτήριο ε, πρωτοτυπίας για κάθε κομμάτι που σου έχει πάρθει από εσένα αν δεν χρησιμοποιήσεις κάποιο λογισμικό ε, τεχνητής νοημοσύνης ε, ιδίως όταν τα αποκόμματα τύπου είναι τόσο μικρά που δεν καλύπτεται το κριτήριο της πρωτοτυπίας. Ωστόσο, αν δείτε όμως ότι υπάρχουν εκατομμύρια τέτοια αποκόμματα, προφανώς η εικόνα αλλάζει. Εκατομμύρια αποκόμματα λοιπόν γίνονται αντικείμενα κλοπής από αυτούς τους aggregator. Όπως λοιπόν οι ε, ε, χίλιες μέλισσες μπορούν να σκοτώσουν έναν άνθρωπο ε, αλλά όχι μία μόνη της έτσι και εκατομμύρια snippets μπορούν να σκοτώσουν έναν εκδότη Ας μην υπάρχουν παρεξηγήσει, λοιπόν, γιατί αυτό είναι μια παρανόηση λόγω του γεγονότος ότι το... δεν έχει αποφανθεί ακόμα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Έχει όμως αποφανθεί το, Ευρωπαϊκό, το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαιο... Ε, δικαστήριο και εκεί ε, το δικαστήριο αυτό ανέφερε και απεφάνθη ότι δεν είναι το ίδιο το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και το δικαίωμα του εκδότη. Το Γερμανικό Ανώτατο Δικαστήριο λοιπόν ε, ξεκαθάρισε ότι αυτά τα ε, συναφή δικαιώματα για δημιουργούς που ε, απολαμβάνουν αυτά τα δικαιώματα υπάρχει παραβίαση ακόμη και αν γίνεται χρήση μόνο μικρών αποσπασμάτων των δημιουργημάτων τους. Γιατί, διότι αυτά τα συναφή δικαιώματα δεν προστατεύουν την πρωτοτυπία αλλά τις επενδύσεις. Και κάθε κομμάτι μιας έκδοσης απολαμβάνει αυτή την προστασία, αυτού του δικαιώματος. Ε, πρόκειται για τις επενδύσεις που κάνουν οι εκδότε, δηλαδή όλε όλες οι επενδύσεις που χρειάζονται για να μπορεί κανεί να συγκεντρώνει και να δημοσιεύει συγκεκριμένο περιεχόμενο. Από αυτή την άποψη πρόκειται για επένδυση και γι' αυτό χέρι της προστασίας νομοθεσία. Τι συμβαίνει σε σχέση με την κατοχή, με την ιδιοκτησία. Αρκεί, όχι. Το να ε, θεωρεί κανείς ότι ε, απολαμβάνει ένα δικαίωμα το οποίο είναι αναποτελεσματικά προφανώς δεν είναι ενδεδειγμένο και δεν αρκεί. Δεύτερον, δεν θα βοηθούσε κάτι τέτοιο, γιατί είναι μια παραδοχή η οποία ε, την οποία μπορεί κανείς να την, ε, να την αντικρούσει. Γιατί οι freelancer, οι ελεύθεροι ε, δημοσιογράφοι, που είναι όλο και περισσότερο, προφανώς δεν θέλουν να μεταφέρουν το δικαίωμα εκπροσώπησής τους στους εκδότες τους. Θέλουν να το διατηρήσουν για τον εαυτό τους. Άρα πρόκειται για εσφαλμένη παραδοχή. Τρίτον, οι εκδότες δεν έχουν κανένα συμφέρον από το να έρθουν σε αντιπαράθεση με τους δημοσιογράφους. Και ένα παράδειγμα είναι ότι το δικαίωμα αυτό το παίρνει από τους δημοσιογράφους η πρόταση και το πάει στου εκδότε. Μα δεν το θέλουν. Οι εκδότε θέλουν οι δημοσιογράφοι να απολαμβάνουν μια ε, συνολικά ε, πιο ισχυρή ε, οικονομία στον τύπο. Δεν θέλουν να έρθουν σε αντιπαραθέσεις με τους δημοσιογράφους του. Παραδείγματα Γερμανία και Ισπανία. Εδώ υπάρχει εσφαλμένη εστίαση. Γιατί μιλάνε όλοι πάντοτε για τον κύκλο εργασιών. Εδώ πρόκειται για δικαίωμα απαγόρευση. Δηλαδή, πλατφόρμες δεν θα μπορούν να εμφανίζονται οπουδήποτε και παντού εκμεταλλευόμενες περιεχόμενο άλλων. Ο βασικός στόχος λοιπόν είναι να μην γίνεται τέτοια εκμετάλλευση από πλατφόρμες. Σκοπός δεν είναι να υπάρχουν, να καταβάλλονται τέλη ε, Αντιθέτως, ε, σκοπός είναι να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των εκδοτών και να μην, δοθεί, να μην δίνονται ε, κίνητρα για να πηγαίνει κανείς και να αντιγράφει τη δουλειά που έχουν κάνει άλλοι και να βγάζει λεφτά με αυτόν τον τρόπο. Δεύτερον, μιλούμε για το δικαίωμα το οποίο έχει θεσπιστεί μόλις εδώ και κάποια χρόνια είναι γνωστό ότι κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχους μηχανισμούς οι οποίοι χρειάζονται χρόνια μέχρι να οριμάσουν. Πρέπει να γίνουν καταγγελίες να να, να, από, από διάφορες πλευρές, να, να αποφανθούν τα δικαστήρια κτλ. κτλ. Μάλιστα στην Ισπανία ε, ακούστηκε ότι οι εκδότες ε, επλήγησαν από αυτό το δικαίωμα. Το αντίθετο συμβαίνει. Πριν από μια εβδομάδα βγήκε μια σχετικά, σχετική μελέτη η οποία απέδειξε ότι η βασική κυκλοφορία, η άμεση κυκλοφορία στις, ε, ε στις εφημερίδες αυξήθηκε στην πραγματικότητα διότι η άμεση χρήση ενός μιας ιστοσελίδας δημιουργεί πιο άμεση χρήση και είναι πολύ πιο πολύτιμη στους εκδότες από ότι το να παίρνεις παραπομπές και links από κάποιες άλλες πλατφόρμες που δεν τις ενδιαφέρει καθόλου το πώς πάει η δική σου εκδοτική επιχείρηση. Γι' αυτό και νομίζω η Γερμανία και η Ισπανία είναι παράδειγμα που μπορεί να, ε, ε, να γίνει αντικείμενο μίμησης. Και αν υπόλοιξαν και κάποιες ελλείψεις και προβλήματα, ε, πεδίο δόξης λαμπρών να τα ξεπεράσουμε. Νομίζω πάντως ότι η Γερμανία και η Ισπανία αποδεικνύουν ότι πρόκειται για μια θετική διαδικασία και όχι το αντίθετο όπως ακούστηκε. Ευχαριστώ πολύ. Τέταρτος και τελευταίος ομιλητής μας είναι ο κύριος Κριστόφ Καρόν που θα παρουσιάσει τις ε, δικές του απόψεις. Έχετε 10 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ σε αυτή την ακρόαση ενώπιον σας. Θα ήθελα να εξετάσω δύο ζητήματα που αφορούν το πολύ ενδιαφέρον ε, θέμα του συγγενικού δικαίου ε, για, τις, ε, για τους ομίλους τύπου. Και το ερώτημα είναι χρειάζεται κάτι τέτοιο. Και το δεύτερο μου ερώτημα είναι ποιο είναι αυτό το ιδανικό συγγενικό δικαίωμα, ποιο θα ήταν το πιο αποτελεσματικό όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, κατά πόσο πρέπει να δημιουργηθεί ένα τέτοιο συγγενικό δικαίωμα για τι επιχειρήσει τύπου, θα σα δώσω μια απάντηση που για μένα είναι προφανή. Η απάντηση είναι καταφατική. Φυσικά και πρέπει να δημιουργηθεί ένα συγγενικό δικαίωμα για την επιχείρηση τύπου. Για ποιο λόγο, διότι μεταξύ όλων των παρόντων όλοι θα συμφωνήσουμε ότι πρέπει να προστατεύσουμε τον τύπο, να τον βοηθήσουμε ο τύπος διαδραματίζει ουσιώδη ρόλο σε μια δημοκρατική κοινωνία, διασφαλίζει την ε, πολυφωνία, ε, είναι, έχει μια αποστολή κοινή ωφελία. Για να προστατεύσουμε λοιπόν τον τύπο πρέπει να του χορηγήσουμε ε, νομικά μέσα που θα τον προστατέψουν. Φυσικά υπάρχει το δικαίωμα του δημιουργού. Το δικαίωμα του δημιουργού είναι αποτελεσματικό σε κάποιο βαθμό. Το αποτέλεσμα δημιουργού προστατεύει τη δημιουργία, τις δημιουργίες που είναι γνήσιες, αυθεντικές. Οπότε υπάρχει ένα αντικείμενο που μας ενδιαφέρει εδώ, αλλά είναι περιορισμένο. Το συγγενικό δικαίωμα προστατεύει την επένδυση. Η επένδυση του τύπου λοιπόν στο νομικό κόσμο είναι κάτι πολύ σημαντικό. Στον κόσμο του πολιτισμού εδώ και 30 χρόνια στον τομέα της μουσικής ε, των οπτικοακουστικών ε, παραγωγών εκεί συχνά υπάρχει ένα δικαίωμα δημιουργού αλλά και ένα συγγενικό δικαίωμα το οποίο αφορά την επένδυση. Για ποιο λόγο? να μην υπάρχει το ίδιο για τις επιχειρήσεις τύπου. Πρέπει να διασφαλίσουμε ίση μεταχείριση μεταξύ εκείνων που επενδύουν και να δώσουμε, να χορηγήσουμε στον τύπο τη δυνατότητα να προστατεύσει τις επενδύσεις με ένα συγγενικό δικαίωμα, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει προκλήσεις ε, στον κόσμο, να καταπολεμήσει αποτελεσματικά την παραποίηση, να αξιοποιήσει τα δικαιώματά της και να καταπολεμήσει το, τα κάποιον τρόπο παράσιτα, τα οποία υποκλέπτουν την αξία που χρησιμοποιεί και χρηματοδοτεί ο τύπος, χωρίς ωστόσο να καταβάλουν οποιοδήποτε τίμημα, δωρεάν, τσάμπα τα παίρνουν όλα αυτά. Κάτι που φυσικά είναι απαράδεκτο. Το δεύτερο θέμα είναι λίγο πιο τεχνικό από νομική άποψη ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός ιδανικού συγγενικού δικαιώματος επιχειρήση τύπου. Μερικές γενικές πληροφορίες πρώτα απ' όλα. Αυτό το συγγενικό δικαίωμα πρέπει να είναι λογικό. Λογικό με ποια έννοια. Πρέπει να επιτυγχάνει μια ε, σωστή ισορροπία μεταξύ τη επένδυσης των επιχειρήσεων τύπου αλλά και τη ελευθερία. Ε, Έκφραση και των λοιπόν θεμελιωδών ελευθεριών. Πιστεύω ότι στο πλαίσιο αυτή τη συζήτηση λοιπόν πρέπει να αποφύγουμε οποιαδήποτε καρικατούρα. Αυτό το συγγενικό δικαίωμα δεν είναι σκιάχτρο. Δεν θέλει να σκοτώσει το δημόσια έκφραση και την ελευθερία έκφραση. Δεν είναι εχθρό. Είναι ένα δικαίωμα το οποίο πολύ απλά θα βοηθήσει τον τύπο να αυτοπροστατευτεί, να αναπτυχθεί στον ψηφιακό κόσμο και να εξελιχθεί για το καλό των πολιτών των καταναλωτών, των ε, ψηφοφόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα δικαίωμα λοιπόν το οποίο θα σέβεται την ελευθερία έκφρασης, θα περιορίζεται χάρη σε διάφορες εξαιρέσεις που προβλέπονται στην πρόταση οδηγίας, αυτό είναι πολύ καλό. Είναι επίσης ένα δικαίωμα το οποίο δεν θα είναι ανώτερο από άλλα δικαιώματα. Στην πραγματικότητα αυτό το συγγενικό δικαίωμα, αυτό το συγγενικό δίκαιο θα έχει την ίδια εμβέλεια με τα συγγενικά δίκαια που υπάρχουν ήδη από το 1992 στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τους παραγωγούς των ε, φωνογραμμάτων, των μαγνητοσκοπήσεων, των εκπομπών, ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο. Αυτό το συγγενικό δίκαιο λοιπόν των άλλων ε, πολιτιστικών παραγωγών στον τομέα των οπτικοακουστικών παραγωγών και της μουσικής είναι κάτι που υπάρχει εδώ και καιρό, λειτουργεί καλά σχετίζεται με το δικαίωμα δημιουργού και το συμπληρώνει και από όσο ξέρω ούτε σκότωσε τη μουσική ούτε τον οπτικό ακουστικό κόσμο, αντιθέτως θα βοήθησε. Μια μικρή διευκρίνηση. Το άρθρο 11 παράγραφος 2 της προτάσης οδηγίας πρέπει να τροποποιηθεί επί του εξή σημείου. Το συγγενικό δικαίωμα της ε, επιχείρησης τύπου δεν πρέπει να είναι κατώτερο από τα συγγενικά δίκαια. Θα πρέπει να είναι ίσο στην ιεραρχία των δικαίων. Αντιθέτως, όσον αφορά τη σχέση του με το δικαίωμα ε, δημιουργού πρέπει να είναι κατώτερο. Γιατί, διότι είναι ένα σημαντικός ε, κανόνας ε, η διανοητική ιδιοκτησία είναι ανώτερο δίκαιο από το συγγενικό δίκαιο. Το συγγενικό δίκαιο αυτό δεν θα ευλάψει τους δημοσιογράφους, δεν θα μπορεί να τους βλάψει, δεν θα μπορεί σε καμία περίπτωση να τους ενοχλήσει. Αντιθέτως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό τώρα, σύμφωνα με τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ του δικαιώματος δημιουργού και των ε, γειτονικών συγγενικών δικαιωμάτων και δικαίων το δίκαιο για τις επιχειρήσεις τι πρέπει να είναι ξεχωριστό από το δικαίωμα δημιουργού. Δεν πρέπει λοιπόν να προστατευθούν οι επιχειρήσεις τύπου επειδή αναγνωρίζουμε ότι ε, περιέχουν γνήσιο περιεχόμενο που προστατεύεται από το δικαίωμα δημιουργού. Πρέπει να προστατεύονται διαφορετικά γιατί ο σκοπό είναι διαφορετικά. Στο δικαίωμα δημιουργού προστατεύουμε το αρχικό δημιούργημα ενώ στο δικαίωμα τη επιχείρηση τύπου ε, προστατεύουμε την επένδυση που μπορεί να αφορά ε, μια εφημερίδα, ό,τι περιλαμβάνει μια εφημερίδα που μπορεί να μην είναι δημιουργία τη ίδια τη εφημερίδα. Ή το απόσπασμα μπορεί να προστατεύεται, το οποίο μπορεί να μην είναι το γνήσιο κείμενο απαραίτητα. Κάτι άλλο σημαντικό σε αυτές τις γενικές μου παρατηρήσεις κατά την άποψή μου είναι σημαντικό που η πρόταση οδηγίας ενδιαφέρεται για το συγγενικό δικαίωμα στον ψηφιακό κόσμο. Αυτό είναι φυσιολογικό. Υποχρεούται κιόλας υποχρεώθηκε και η οδηγία για το δικαίωμα δημιουργού να ασχοληθεί με τον ψηφιακό κόσμο. Αλλά το σημαντικό είναι ότι αυτή η πρόταση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμποδίσει τα κράτη-μέλη από το να δημιουργήσουν ένα συγγενικό δίκαιο που να υποστηρίζει ε, τις επιχειρήσεις τύπου και για τον έντυπο τύπο. Διότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, το βρίσκουμε σε πολλέ αποφάσει του δικαστηρίου. Ε, αυτή την αρχή τη τεχνολογική ουδετερότητα. Δεν θα κάνουμε απαραίτητα διάκριση ανάλογα με το αν η εκμετάλλευση γίνεται στον ψηφιακό κόσμο ή στον αναλογικό κόσμο. Και αυτό θα ήταν ενδιαφέρον λοιπόν να αφήσουμε τα κράτη-μέλη ελεύθερα όταν θα μεταφέρουν το δίκαιο αυτό, εφόσον θα υπάρξει το δικαίωμα, το δικαίωμα αυτό, να του δώσουμε τη δυνατότητα να ε, προστατεύουν ε, και το δικαίωμα αυτό στον ε, κόσμο, στο μη ψηφιακό κόσμο. Τώρα κάποια νομικά ζητήματα, το αντικείμενο του δικαίου, όπω ορίζεται στο άρθρο 2.4 τη πρόταση οδηγία, εμένα μου φαίνεται τέλειο. Πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ σαφέ και μάλιστα αναφέρουμε όλα τα μέσα. Κάτι που υπενήστε ότι τύπος δεν είναι μόνο ε, ο ψηφιακός κόσμος. Ε, για μένα λοιπόν ε, είναι πάρα πολύ καλό αυτό που αναφέρεται στο 2.4 αλλά θα πρέπει να προβληματιστούμε κατά πόσο θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τα πρακτορία τύπου στο πλαίσιο αυτού του συγγενικού δικαιώματο, του συγγενικού δικαίου, γιατί και αυτέ κάνουν επενδύσει και αυτέ έχουν δημοσιογράφου και δημοσιογραφική παραγωγή. Ε, έχουν και δραστηριότητε εμπορικέ στι ε, ιστοσελίδε του. Και αυτό πιστεύω ότι θα έχει κάποιο ενδιαφέρον. Τώρα, όσον αφορά το περιεχόμενο του δικαίου αυτού, του δικαιώματο αυτού, θα πρέπει να είναι συγγενικό, αποκλειστικό δικαίωμα άδεια ή απαγόρευση το να δημιουργηθεί ένα τεκμήριο αντιπροσώπευσης του δικαιώματο δημιουργού είναι περιττό ω πρόταση. Δεν ε, εξυπηρετεί κανένα σκοπό, είναι αναποτελεσματική και περιπλέκει χωρί λόγο τι σχέσει μεταξύ των επιχειρήσεων που απασχολούν ε, με, τους και του δημοσιογράφου που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Ε, στη Γαλλία α πούμε με μια τέλεια νομοθεσία από το 2009. Ειλικρινά καλύτερα να μην κάνουμε τίποτα παρά να δημιουργήσουμε αυτού του είδους το τεκμήριο αντιπροσώπευσης το οποίο θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στην αστική δικονομία και στο δικαίωμα στο ενοχικό δικαίωμα, στο δίκαιο. Όπως και στις, στις επιχειρήσεις τύπου λοιπόν, όπως και στα συγγενικά δικαιώματα θα πρέπει να γίνεται αναφορά στην πρόταση οδηγία στην οδηγία 2006-615 ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε οι επιχειρήσεις τύπου να χαίρουν και ενό δικαιώματος διανομής ε, το οποίο μπορεί να έχει μια χρησιμοποίηση. Τώρα όσον αφορά τα τα αποσπάσματα, η πρότασή μου είναι η εξή. Ο νόμος, η οδηγία, κυρίως στον τομέα της τεχνολογίας, πρέπει να θεσπίζει κάποιες ε, γενικές, ε, αρκετά ευρείες αρχές ε, για να προλάβει τις εξελίξεις στο μέλλον χωρίς να απαρχιωθεί γρήγορα. Δεν απαιτείται να αναφέρουμε ρητά τα snippet. Σήμερα μιλάμε για snippet, σε πέντε χρόνια θα μιλάμε για κάτι άλλο. Αυτό που χρειάζεται είναι κάποιο μονοπόλιο, αρκετά γενικόλογο, ώστε να παραμείνει επίκαιρο μέσα στο χρόνο. Και μετά η νομολογία, το δικαστήριο, οι εθνικοί δικαστέ θα καθορίζουν κατά περίπτωση κατά πόσο τα αποσπάσματα θα περιλαμβάνονται ή όχι στο μονοπόλιο. Το ίδιο και για τα υπερκείμενα, για τα hypertext. Ε, εκεί μπορούμε να κάνουμε τεράστιε συζητήσει, αλλά δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε σαν είναι κάτι ιδιαίτερο στον τύπο. Είναι κάτι που ε, αφορά όλο το δικαίωμα δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα. Ε, αναφέρεται σε αυτό το δικαστήριο. Σα ελπίσουμε λοιπόν ότι απλά το δικαστήριο θα εξελίξει κάποια νομολογία του όταν μιλάμε τώρα για κερδοσκοπική χρήση, κερδοφόρο χρήση υπερσυνδέσεων για αποκόμιση χρηματικού κέρδους. Τώρα, η 20 ετής προστασία, πριν τελειώσω γιατί όχι, δεν είναι καν πολύ. Δεν είναι αρκετός χρόνος, δεν επιτρέπει ε, στις επιχειρήσεις ε, τύπου να προστατεύσουν τα, και να αξιοποιήσουν τα αρχεία τους ε. Ε, γιατί έχει 50 χρόνια. Και τέλο, θα πρέπει να καλύψουμε οπωσδήποτε ένα κενό που υπάρχει στην πρόταση οδηγία. Πρέπει οπωσδήποτε να δώσουμε στι επιχειρήσει τύπου τα μέσα να καταπολεμήσουν την παραποίηση. αναφερόμενη στην οδηγία 2004-48 που αφορά την υπεράσπιση τη διανοητική ιδιοκτησία. Εγώ εκφράζω την επιθυμία το κοινοβούλιο σα να δώσει τα ένδικα μέσα ε, στην ε, ε, σε επιχειρήσεις τύπου για να αναπτυχθούν στον ψηφιακό κόσμο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς ευχαριστούμε λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα έχουμε ερωτήσεις από πλευρά των συναδέλφων και στη συνέχεια θα μπορέσετε να δώσετε απαντήσεις αν θέλετε. Ο κύριος Καβαντάκης ζητήσει πάντως το λόγο. Ευχαριστώ και εσάς Πρόεδρε και τους ε, ομιλητές μας. Μας είπαν τις απόψεις τους που είναι διαφορετικές και ε, όλα αυτά είναι ε, αποτέλεσμα καθαρά διανοητικής προσπάθειας και δεν πρόκειται για αποτέλεσμα επιρροής, κάτι το οποίο το γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει. Τώρα να δούμε τι γίνεται όσον αφορά κάποια πολιτική αποτίμηση του θέματος και βέβαια εδώ έχουμε και διαφορετικές κομματικέ τοποθετήσει και έχουμε κάποιο είδου ε, που ισχύει σχετικά ε, για παράδειγμα αυτοί που προσπαθούν να εντάξουν την Ευρώπη σε ένα πλαίσιο υποταγής θα έλεγα υποταγής σε κάποια τεχνολογία που έτσι κι δεν την έχουμε οπότε έπρεπε όλη η νυφάλια να κάτσουμε και να σκεφτούμε επί τη βάση ιδεών και αρχών ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει αυτές να τις υπερασπίζει γιατί είναι αυτές τα θεμέλια του πολιτικού διαλόγου που ήδη αρκετά <clears throat> ταλαιπωρείται σήμερα από το χρήμα και από τους εξτρεμιστές. Άρα εμείς θα πρέπει να λάβουμε τις ευθύνες μας, τόσο ώστε να υπάρχει αυθεντικά η έννοια του δημιουργού και έτσι εμεί να κάτσουμε και να νομοθετήσουμε για να θεσπίσουμε ένα θηγείο ε, χωρίς ε, να μπορούμε να ρυθμίσουμε κάθε λεπτομέρεια γιατί οι λεπτομέρειες ε, εξελίσσονται οπότε κανείς θα πρέπει συνεχώς να διορθώνει την νομοθεσία αλλά θα πρέπει να χαράξουμε και τον στόχο όλων αυτών ο στόχος αν μου επιτρέπετε ε, νομίζω ότι ορίζεται από δύο διαπιστώσεις και συχνά έχουμε πει ότι οι Ευρωπαίοι ε, είμαστε σαν τις χώρες του κόλπου μεταξύ των δύο πολέμων γιατί έχουμε πολύ πετρόλαιο δηλαδή την παραγωγή του περιεχομένου και ο πολιτισμός των 28-27 σε λίγο είναι μια στήρευτη πηγή τέτοιου περιεχομένου αλλά δεν έχουμε όπως τότε οι χώρε του κόλπου και οι χώρε που έχουν το φυσικό δεν έχουμε τα μέσα εξόριξης ούτε να μεταφέρουμε το πετρέλαιο ούτε να έχουμε κάποιο είδους δηληστήρια ούτε μπορούμε και να κάνουμε τη διανομή γιατί έχουν στα, στα χέρια των Αμερικανών τα μέσα ή Ασιατών Κινέζων ουσιαστικά επομένως το δημοκρατικό μας καθήκον είναι ακριβώς το πώς θα προστατεύσουμε αυτό το περιεχόμενο. Δεν είναι θέμα ε, business, δεν είναι επιχειρηματικό, δεν είναι θέμα lobbying και επιρροής. Είναι κάτι ε, για το οποίο θα πρέπει να δώσουμε λόγο για να το καταφέρουμε. Να προστατεύσουμε, να αξιοποιήσουμε και ε, αυτοί οι οποίοι θέτουν αυτό το περιεχόμενο σε εμπορία θα πρέπει να αμείβονται. Αυτό με ενδιαφέρει και τώρα αυτό με οδηγεί σε μια άλλη σκέψη. Ότι Πρόκειται για κάποιες ιδέες που είναι δυναμικές, ε, μη μια ατμομηχανή εδώ πέρα στην ειρηνική ήπειρό μας που καμιά φορά διακόπτει η ειρηνική πορεία δυστυχώς από πολέμους οπότε καθήκον μας είναι να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε αυτό το τα περιεχόμενα στην υπηρεσία της δημοκρατίας ε, χωρίς αυτό να μας οδηγεί σε κάποιο είδου υποδούλωση ε, και ειδωλολατρεία. Επομένως χρειάζεται κάποιο είδους ε, υγιής ρύθμιση, ελευθερία ε, και απλώς ιδεολογικής. Δεν μπορεί να έχουμε άλλου είδους βάση επιχειρηματολογίας. Πέραν αυτόν τώρα, να δούμε από πλευράς του πολίτη που έχει επίγνωση του καθηκοντός του. Θα πρέπει από εδώ να δούμε τι οικονομικά ζητήματα γεννώνται και τι επίσης ε, ισχύει νομικά μετά από όλα όσα ακούσαμε. Γι' αυτό σας λέω ότι με βάση όλα αυτά θα πρέπει, κυρίες και κύριοι, πρόεδρε, θα πρέπει κάθετα να είμαστε κατά μια ιδέα που κυκλοφορεί στην Ευρώπη. Είναι κάποιο είδου ε, πρόταση ανοχής και ανεκτικότητας, γιατί όταν μιλούμε για περιεχόμενο, μιλούμε για κάποιους οι οποίοι επιζούν με αυτά τα οποία δημοσιεύουν και παράγουν. Ιδάλλως, τι είναι, είναι, σαν έμποροι πορτοκαλιών, ποδηλάτων, ρούχων. Οπότε θα πρέπει να γράψουμε δύο λέξεις νομικές και να πούμε ότι μπορεί κανείς να πουλήσει κάτι που δεν έχει αγοράσει. Πώς θα το πούμε αυτό. Άρα θα πρέπει να βγούμε από αυτή την επιχειρηματολογία δηλαδή όσον αφορά αυτή του είδους τη θέση σε εμπορία και την αγορά και να δούμε πώς θα αγκαλιάσουμε, πώς θα συνεχίσουμε αυτό που είπανε δύο τουλάχιστον τους ότι δηλαδή ο στόχος είναι να έχουμε ένα πλαίσιο σύμφωνα το οποίο οι επιχειρήσεις να μπορούν να είναι ελεύθερες από πλευρά οικονομικής και ιδεολογικής και σας ευχαριστώ και θα πρέπει να μιλήσουν και οι άλλοι συνάδελφοι. Ευχαριστούμε κύριε Φως, ο εισηγητής μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους ομιλητές για τις παρουσιάσεις τους. Αυτό που κατά τη γνώμη μου δεν φωτίστηκε παρακώς είναι η σημασία που έχει η ύπαρξη μιας ελεύθερης, ανεξάρτητης ε, ε, ε, του ελεύθερου και του ανεξάρτητου τύπου για το δημοκρατικό μας πολίτευμα. Έχουμε λοιπόν μια συζήτηση για την πολυφωνία, τον πλουραλισμό, την, τη λειτουργία του, του δημοκρατικού συστήματος. Γι' αυτό και ο δημοκρατικός και ανεξάρτητος τύπος αποτελεί πυλώνα του δημοκρατικού πολιτεύματος. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι ποιος είναι ο ρόλος του τύπου και ποια, είναι η σημασία που έχει ο τύπος για τις κοινωνίες μας. Και εδώ η απάντηση είναι προφανής. Ο τύπος είναι σημαντικός, είναι αναγκαίος και γι' αυτό πρέπει να στείλουμε ένα στεναρό μήνυμα και να πούμε ότι έτσι όπως γίνονται τα πράγματα μέχρι τώρα δεν μπορούν να συνεχίσουν. Και νομίζω ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο να πει κανείς ναι, άλλαξαν οι συμπεριφορές των χρηστών και έτσι μειώθηκαν οι, τα έσοδα. Και άλλο πράγμα να πει κανείς ότι η εμπορία και εκμετάλλευση περιεχομένου χωρίς κανόνες από τον καθένα όπως νομίζει και όπως θέλει. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Στο κρατήριο από το οποίο κατάγομαι, κατάγομαι εγώ γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια μια αξιολόγηση, ένας απολογισμός του τι γίνεται ε, στην, ε, ε, στον τομέα του τύπου, στον κλάδο του τύπου. Μάλιστα, η τελευταία σχετική έκθεση, η οποία συντάχθηκε και υπό κυβέρνηση σοσιαλδημοκρατών και πρασίνων, περιέχει στοιχεία που είναι τουλάχιστον ανησυχητικά, για να μην πω τρομακτικά. Μειώνονται τα έσοδα, μειώνεται η ποιότητα. Η κυβέρνηση ε, του κρατηδίου ε, θέλει να εξασφαλίσει τα δικαιώματα των εκδοτών και των ε, δημιουργών. Αν δει όμως κανείς πόσο έχει μειωθεί η πολυμορφία και η πολυγλωσία και η πολυφωνία, με συγχωρείτε, στον τύπο, μπορεί να μην είναι ακόμα ζήτημα ζωής και θανάτου, για τον τύπο, αλλά είναι σίγουρα ένα σήμα ότι κάτι πρέπει να γίνει και μάλιστα σχετικά άμεσα, ώστε να μπορεί ο τύπος να επιτελεί το έργο του, να επιτελεί την, την κοινωνική του, τον κοινωνικό του ρόλο, τον δημοκρατικό του ρόλο. Το να μπορούμε δηλαδή μέσω του, της, ε, της πολυφωνίας, του, του πλουραλισμού να εξασφαλίζουμε την ε, ενημέρωση Ιδίω σε μια εποχή των ψευδών ειδήσεων, των fake news, ε, είναι όλα αυτά στοιχεία που μας δείχνουν πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μια υψηλή ποιότητα δημοσιογραφία. Προφανώς τα πράγματα δεν μπορούν να μείνουν έτσι όπως είναι σήμερα και αν τα δει κανεί και διαβαθμισμένα θα μπορούσε ενδεχομένως ε, ακόμη και να θεσπιστεί υποχρέωση αμοιβή αλλά δεν πάει μέχρι εκεί η πρόταση. Δεν, έχει, δεν περιλαμβάνει κάτι τέτοιο ακόμα η πρόταση. Αν δει όμως κανείς ποιο θα είναι το επόμενο βήμα, σε περίπτωση που τα αφήσουμε έτσι όπως έχουν τα πράγματα, τότε αναρωτιέμαι, αυτό είναι πραγματικά το σταθερό, το στεναρό μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε σε όλες τις πλευρές και το οποίο είναι ότι για εμάς ο ελεύθερος και ανεξάρτητος τύπος έχει ε, σημαντικότατο ρόλο να επιτελέσει ακόμη και συνταγματικά. Και αν, ε, αν, αν κοιτάξω λοιπόν αυτή την, ε, το, το συγγενικό ε, δικαίωμα, το συγγενικό δίκαιο που εσείς από ό,τι κατάλαβα προτιμάτε, αυτό είναι το μέλλον δηλαδή του τύπου, εγώ θα έλεγα όχι. Διότι αφού αν παραμείνουν τα πράγματα όπως έχουν, θα πρέπει κάθε φορά, κάθε δημιουργός να αποδεικνύει το ύψος και το επίπεδο της δικής του δημιουργίας. Γι' αυτό και δεν, μπορώ, δεν θεωρώ ότι ε, το να, θα είναι επαρκές το μήνυμα ε, στις πλατφόρμες και στους news aggregators αν τους πούμε ότι απλά θα συνεχίσουμε όπως ε, ε κάναμε μέχρι σήμερα. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια στεναρή, μια σοβαρή παρέμβαση στην, πραγματικό, στην πράξη, ε, σε αυτό που ισχύει σήμερα και μάλιστα χωρίς καν να θεσπίσουμε υποχρέωση αμοιβή. Όχι αντίθετα, θεσπίζουμε νομοθεσία η οποία από μόνη της δεν παράγει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αντιθέτως, κάθε ε, εκδοτικός οίκος, κάθε ε, επιχείρηση του τύπου θα αποφασίσει πώς θα εφαρμόσει την νομοθεσία αυτή με τις δυνατότητες που τις ε, αφήνει βεβαίως εντός των πλασίων της εννοείται. Αλλά αυτό είναι πάλι πολύ διαφορετικό από αυτό που υπόθηκε ότι προτείνεται. Αν λοιπόν σταθμίσουμε τη σημασία της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας από τις μεγάλες πλατφόρμες και ενός δικαιώματος και, και ένα δικαίωμα να μείνονται κατά της κλοπής του περιεχομένου τους, εγώ βεβαίως δεν μπορώ παρά να οδηγηθώ στο συμπέρασμα ότι πρέπει να εξασφαλίζεται δίκαιη αμοιβή των εκδετών. Φυσικά μπορεί κανείς να πει ότι το, το δίκαιο υπερπροστασίας της πνευματικής ε, ε ιδιοκτησίας Μπορεί να μην είναι από μόνο του επαρκέ, αλλά να σας πω την αλήθεια μέχρι στιγμής δεν έχω ε, ακούσει και καμιά άλλη ιδέα για το πώς μπορούν να προστατευτούν τα δικαιώματα των ε, δημιουργών. Βεβαίως, όλοι συμφωνούμε ότι η ανεξαρτησία του τύπου πρέπει να προστατεύεται και να εξασφαλίζεται και δεν πρέπει να, κάνουμε, ε, να, να φανούμε αδύναμοι σε αυτό το μέτωπο. Βεβαίω, προκύπτουν και μια σειρά από ερωτήματα. Αφενός, Συμμερίζεστε την άποψή μου ότι ο τύπος εξακολουθεί να έχει κάποια αξία και για την κοινωνία και τη λειτουργία της. Ότι δεν είναι απλά μια επιχείρηση, δηλαδή μια, μια επιχείρηση του τύπου που απλά βγάζει χρήματα. Δεύτερον, έχετε την αίσθηση ότι οι εκδοτικοί οίκοι και οι δημοσιογράφοι πράγματι αμείβονται ε, δίκαια ε, έχοντας κατά νου αυτά που κάνουν οι πλατφόρμες. Μάλιστα ακούστηκε ότι η κατάσταση στη Γερμανία και στην Ισπανία δεν αρκεί. Ε, υπάρχουν, υπάρχει το πρόβλημα με τα snippets και τα links και τα αποκόμματα. Εγώ να σας πω την αλήθεια δεν παρατήρησα πουθενά ε, να μειώνεται ο αριθμός των links και των snippets λόγω αυτής της νομοθεσίας εκεί όπου θεσπίστηκε. Αλλά επειδή είμαι νομικός πρέπει να σας πω ακόμη και αν διαπιστώσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, είμαστε βέβαιοι ότι όλα αυτά μπορούν να ρυθμιστούν και να διευθετηθούν νομικά. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς την ίδια άποψη. Επίσης, μιλήσατε για δημοσιογράφους που δεν θέλουν το δικαίωμα αυτό, καθώς και εκδόσεις που δεν θέλουν το δικαίωμα αυτό. Εγώ μιλώντα με την, με την Ομοσπονδία, με την Ευρωπαϊκή αλλά και τη Γερμανική Ομοσπονδία ε, εκδοτών έχω αντίθετη άποψη, αντίθετη γνώμα. Αρχικώ πράγματι είχαν διαφωνίε, αλλά πλέον θέλουν ε, να θεσπιστεί ένα τέτοιο δικαίωμα βεβαίως και με συμμετοχή ε, των δημοσιογράφων. Και αυτή η συμμετοχή μάλιστα μπορεί και να ρυθμιστεί νομοθετικά. Επίσης, τι γίνεται αν οι εκδότες δεν θέλουν. Μα δεν είναι υποχρεωμένοι άλλωστε να κάνουν χρήση αυτής της νομοθεσίας. Στις ΗΠΑ όμως υπάρχει και μια κίνηση ε, σύσταση κοινοπραξιών από μικρούς εκδότες ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν την εξουσία και τη δύναμη των μεγάλων πλατφορμών. Άρα η σύστασή μου είναι εκδότες να συστήσουν κοινοπραξίε, να, αναλάβουν κοινέ πρωτοβουλίες ώστε να μπορούν να διαπραγματεύονται επί ίσης με τις πλατφόρμες. Με άλλα λόγια δηλαδή, δεν θεωρώ ότι οι εξελίξεις, αν δεν παρέμβουμε ή αν πούμε απλά ότι θα κάνουμε απλά κάποιες διακοσμητικές αλλαγέ, ότι θα αυτορυθμιστεί. Δεν το πιστεύω αυτό. Αν κάποιος είχε ασχοληθεί με το θέμα σε βάθος από την αρχή, τότε ενδεχομένως να μην ήμασταν καν εδώ και να μην συζητούσαμε τα θέματα που συζητούμε. Αλλά επειδή τα πράγματα ήρθαν στο σημείο που, στο οποίο έχουν πλέον φτάσει, δεν αρκούν κάποιες διακοσμητικές επιμέρους αλλαγές και τροποποιήσεις. Αν θέλουμε δηλαδή πραγματικά να διατηρηθεί ο ανεξάρτητος και ελεύθερος τύπος. Γι' αυτό και θα ήθελα τη δική σας εκτίμηση. Ποια είναι η κατάσταση στον τύπο. Αν η καινοτομία με τα, links και, με την, και, και αν υπάρχει δικαιότερη αμοιβή ε, και αποζημίωση πλέον ε, στην Ισπανία και στη Γερμανία χάρη στην ε, θέσπιση αυτού του δικαίου. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε ένα μικρό χρονικό προσδιορισμό, περιορισμό, συγγνώμη. Έχουμε, έχουμε μόλις 20 λεπτά. Οπότε παρακαλώ, όταν παίρνετε το λόγο, έχετε υπόψη ότι αν θέλετε να ακούσετε και τις απαντήσεις των ομιλητών μας, θα πρέπει κάπως να είστε σύντομοι για να προλάβουμε στο χρόνο που έχουμε διαθέσιμο για το εργαστήριο αυτό. Η κυρία Ράιντερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον καθηγητή Μπέντλεϊ όσον αφορά τα hyperlinks. Αν σας κατάλαβα καλά, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, δεν είπατε ότι το συγγενικό δικαίωμα και το, το δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας έχουν το ίδιο αντικείμενο. Το αφήσατε ανοιχτό και προσωπικά πρέπει να πω ότι συμφωνώ με την ερμηνεία του καθηγητή Χέπνερ ότι το ε, συγγενικό δικαίωμα είναι ευρύτερο από το ε, δικαίωμα διανοητική διαδιοκτησίας και εκεί είναι ακριβώ το θέμα. Νομίζω ότι ο καθηγητής Χεπνερ είπε κάτι πολύ ενδιαφέρον ότι σκοπός του συγγενικού δικαιώματος είναι η απαγόρευση ώστε να διασφαλίσει ότι οι επιχειρήσει που συνδέονται με τους εκδότες δεν θα υπάρχουν και μετά από την εισαγωγή του συγγενικού δικαιώματος υπάρχει λιγότερη κίνηση παραπομπής. Η κίνηση παραπομπής είναι αυτή που ουσιαστικά τα δημιουργείται όλα αυτά. Οπότε αν υπάρχουν λιγότερες παραπομπές αυτό σημαίνει ότι λιγότερος κόσμος έχει κάνει κλικ σε υπερσυνδέσεις. Και το ερώτημα μου είναι αν εσείς εμένετε στη μελέτη σας ότι τα hyperlinks θα επηρεαστούν από αυτή τη νέα πρόταση διότι όπως είπατε ακόμα και το κείμενο του hyperlink μπορεί να θεωρηθεί παραβίαση. Και όπως γνωρίζετε πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν θέσει αυτό το θέμα ότι το συγγενικό δικαίωμα θα επηρεάσει αρνητικά τα hyperlinks. Τι λέτε στους ισχυρισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι αυτό το ενδεχόμενο είναι αδύνατο απλά και μόνο διότι υπάρχει μια αιτιολογική σκέψη που λέει ότι κάθε φορά που δεν κοινοποιείται ένα hyperlink στο κοινό τότε δεν επηρεάζεται από το δικαίωμα. Διότι εγώ από τι εξηγήσει που άκουσα από τον κύριο Χαπνέρ μου κατέστη απολύτω σαφές ότι το να απαγορεύσουμε το linking είναι ακριβώ ο λόγο για τον οποίο ζητούν αυτό το συγγενικό δικαίωμα οι εκδότε, Γιατί φυσικά αν υπάρχει περισσότερη απευθεία κίνηση το κόσμο πάει ε, στις ιστοσελίδες των εκδοτών που ήδη γνωρίζουν που είναι μεγάλοι εκδότε. και μου φαίνεται πολύ δροσιστικό να το ακούω αυτό από κάποιον ε, τον οποίο κανένα δεν θα υποψιαστεί ότι υποστηρίζει του μεγάλου επιχειρηματίε, ότι σκοπό του γειτονικού δικαιώματο δεν είναι να πληρώσει το Google και το Facebook και οι λοιπέ εταιρείε, αλλά απλά να απογορεύσει την κίνηση μέσω παραπομπών, που είναι το hyperlinking. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριο Άντρεσον. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, πιστεύω ότι αν θέλουμε καλά μέσα και ανεξάρτητα θα πρέπει να υπάρξει τεράστια δημόσια χρηματοδότηση, η οποία φυσικά θα πρέπει να γίνει από τα κράτη-μέλη. Και χαίρομαι λοιπόν που ακούω όλα αυτά τα όμορφα λόγια για το πόσο σημαντικά είναι τα ελεύθερα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ναι, ξέρετε κάτι, πρέπει να κινητοποιήσουμε πόρους και αυτό πρέπει να γίνει με δημόσιο χρήμα. Ήθελα να ρωτήσω τους συντάκτες των μελετών τι ποσά μπορούμε να κινητοποιήσουμε μέσω αυτής της πρότασης όπως το καταλαβαίνω εγώ, μιλάμε για μικρά ποσά σε σχέση με αυτά που θα χρειαστεί ο ελεύθερος τύπος για να μπορέσει να παραδώσει δημοσιογραφία υψηλού επέδου και υψηλής ποιότητας ισχύει αυτό. Ευχαριστώ κύριε Ζεύκα. Ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό ακριβώς ήθελα να αναφερθώ στα όσα είπε μόλις ο κύριος Άντερσον Μιλάμε για τη δημοσιογραφία υψηλή ποιότητα. Πρώτα απ' όλα, η κατασκευή αυτού του δικτύου δημοσιογραφία υψηλή ποιότητα και η διατήρηση αυτού του δικτύου απαιτεί τεράστιε επενδύσει. Αυτό ανεξάρτητα από τον δημόσιο ιδιωτικό χαρακτήρα των ε, εν λόγω μέσων. Εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τα αποτελέσματα που θα θέλουμε να έχουμε στην αγορά. Και ό,τι και να πούμε εδώ για τα συγγενικά δικαιώματα, των οποίων δικαιούχοι είναι οι, οι, εκδότες ε, τύπου. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι τα δικαιώματα αυτά ε, δεν θα εξυπηρετήσουν μόνο τους μεγάλους, αλλά όλο τον κόσμο. Ανεξαρτήτως μεγέθους των επιχειρήσεων αυτών, η κάθε επιχείρηση έχει κάποιο συγκεκριμένο συμφέρον και έχει κάποιο αναγνωστικό κοινό το οποίο θα πάει να αναζητήσει τι πληροφορίε που παρέχει η συγκεκριμένη επιχείρηση ξέροντα ότι αυτέ τι πληροφορίε είναι καλέ, αληθεί, επαληθευμένε. Οπότε ο αναγνώστης πάει μόνο του να ψάξει να βρει τον τοπικό ε, εκδότη ή μια μεγάλη επιχείρηση. Δεύτερη ερώτηση. Αυτό το hyperlinking είναι η σύνδεση μεταξύ των εκδοτικών οίκων και των μεγάλων πλατφορμών. Ποιος απαγορεύει σε αυτές τις μεγάλες πλατφόρμες online και αυτές να είναι επιχειρήσεις ενημέρωσης, επιχειρήσεις τύπου. Εάν το επιθυμούν, ποιος φέρει το κόστος, ποιος επενδύει για αυτές τις υποδομές που επιτρέπουν την παραγωγή περιεχομένου, δημοσιογραφικού υψηλού περιεχομένου. Εάν το μάθουμε αυτό, εάν ξέρουμε ποιο πραγματοποιεί αυτές τις επενδύσεις, τότε θα μπορούμε να μιλάμε για ίδιους κανόνες. Αλλιώς πρόκειται για Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν μπορώ να δώσω το λόγο αυτή τη στιγμή στον κύριο Αριμό, διότι θα ήταν κατά, τον, κατά του κανονισμού. Αν προλάβουμε αργότερα, τότε θα δούμε. Δίνω το λόγο τώρα στην Κομισιόν, στον κύριο Αμπραμόντε. Για μια σύντομη αντίδραση. <laughs> <laughs> Λοιπόν, πολύ γρήγορα για τη μελέτη θα πρέπει να μην εξάγουμε τεράστια και οριστικά συμπεράσματα από μια μελέτη τόσο περιορισμένου εύρους. Λίγες αναθεωρήσεις, ε, εννιά ερωτηθέντες, δεν είναι πολύ σημαντικό το δείγμα. Στόχος της μεταρρύθμισης, ένας από τους βασικούς ε, στόχους της μεταρρύθμισης ε, του δικαιώματο της διανοητικής ιδιοκτησίας είναι να παρέχουμε ίσους κανόνες στο παιχνίδι ώστε όλοι να μπορούν ε, να έχουν έλεγχο και να παρακολουθεί το περιεχόμενο που χρησιμοποιούν τα τρίτα μέρη. Αυτό ενισχύει τη θέση των εκδοτών ενώπιον των πλατφορμών οι βγάζουν χρήματα με το περιεχόμενο που δημιουργούν οι εκδότες. Υποστηρίζοντας τους εκδότες και το σχετικό τομέα, όπως υπόθηκε πολύ όμορφα από τον κύριο Βος, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας ε, του τύπου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα επηρεάσει θετικά την ποιοτική δημοσιογραφία. Πιο συγκεκριμένα θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε το τρομακτικό φαινόμενο των ε, fake news, των ψευδών Κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι η πιο αντιπροσωπευτική ομοσπονδία δημοσιογραφών σε μια επιστολή της ε, προς ε, την Κομισιόν, η EFJ, επεσήμανε αυτό το σημείο και είπε ότι είναι έτοιμη να υποστηρίξει την πρόταση της Κομισιόν ακόμη και να πάει παραπέρα βελτιώνοντας την ε, εφαρμογή του δικαιώματος ε, των ε, εκδοτών τύπου. Τώρα για το πεδίο εφαρμογής και τα αποτελέσματα. Πιστεύω προσωπικά ότι η κίνδυνη που επισημαίνει η μελέτη είναι λίγο υπερβολική. Επίσης δεν συμφωνώ απόλυτα με τον καθηγητή Χόπνερ όσον αφορά το πεδίο των δικαιωμάτων. Στην αιτιολογική σκέψη 34 λέμε σαφω ότι τα δικαιώματα που χορηγούνται στους εκδότε δημοσιευμάτων τύπου ε, στο πλαίσιο αυτή τη οδηγία, θα πρέπει να έχουν το ίδιο πεδίο εφαρμογή ε, όπως και για την αναπαραγωγή και τη διάθεση στο κοινό όσον αφορά την ψηφιακή χρήση. Ουσιαστικά το πεδίο εφαρμογή του νέου δικαιώματο και του γειτονικού δικαιώματο και το πεδίο εφαρμογή του δικαιώματο τη διανοητικής διεκτησία συμπίπτουν. Οπότε εδώ δεν αλλάζουμε το πεδίο εφαρμογή το αντικείμενο. Οπότε οι καταναλωτές, οι πολίτες, οι ιδιώτες θα μπορούν με τους ίδιους περιορισμούς να μοιράζονται snippets και hyperlinks. Όπως κάνουν και σήμερα. Με άλλα λόγια, πιστεύουμε ότι το συγγενικό δικαίωμα δεν θα κάνει τα πράγματα χειρότερα για τους καταναλωτές, για τον πολίτη. Το ίδιο ισχύει και αυτό δεν έχει συζητηθεί. Το ίδιο ισχύει λοιπόν και για τις εξαιρέσεις. Τις ίδιες εξαιρέσεις που έχουμε για το copyright και ειδικότερα η εξαίρεση της παράθεσης, του quotation exception και αυτό θα ισχύει ε, και στο συγγενικό δικαίωμα. Οπότε είναι σημαντικό να μην υπερβάλλουμε ε, ποιες θα είναι οι αθέλητες ε, συνέπειες της πρότασης επί της ελευθερίας του λόγου και για τους πολίτες. Δύο ακόμα σημεία μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά τις διαφορές μεταξύ της γερμανικής και ισπανικής νομοθεσίας ε, και ε, της πρότασης αυτής, πιστεύω ότι η μελέτη έπρεπε να αφιερωθεί λίγο περισσότερο ε, στις διαφορές. Πρώτα απ' όλα, δεν απαιτούμε από τους εκδότες να απαιτούν αποζημίωση. Δεν υπάρχει υποχρέωση απέτηση αποζημίωση, αντίθετα με το ισπανικό σύστημα, δεν υποχρεούμε συλλογική διαχείριση. Υπάρχει μια βασικότατη διαφορά επίση, πιστεύω, σαν αυτή, αλλά κάτι πιο σημαντικό είναι ότι ακολουθούμε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση που θα είναι το αντίθετο, το αντίστροφο του κατακαιρματισμού. Ένα άλλο σημείο το οποίο έχουμε παραβλέψει, ε, τη διαφάνεια και τους μηχανισμούς προσαρμογής της αποζημίωσης προς όφελος των δημιουργών και των ε, ερμηνευτών. Ε, χαιρόμαστε με αυτά προτείνονται στην πρόταση Τη Κομισιόν, αλλά δεν καταλαβαίνουμε γιατί θα έπρεπε να είναι πιο φιλόδοξη. Τι δεν λέμε δηλαδή. Τι δεν λέτε στη μελέτη σας. Κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι εμείς πιστεύουμε πω συνολικά η διαφάνεια στις συμβάσει και στους συμβατικούς μηχανισμούς θα λειτουργήσει προ όφελο των δημιουργών και των ερμηνευτών στην Ευρώπη. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα από τη μελέτη σα λέτε ότι στη Γερμανία δεν υπάρχει γενικό ε, εναλλακτικό σύστημα επίλυσης διαφορών προς όφελος των δημιουργών. Ε, αυτό θα δημιουργήσουμε και εδώ. Ένα εναλλακτικό ADR για τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές. Ως αποτέλεσμα της πρότασης αυτής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Και τώρα, στο πιο δύσκολο φτάσαμε όσον αφορά τους καλεσμένους μας. Έχει ο καθένας από εκείνους δύο λεπτά για να απαντήσει. Ας ξεκινήσουμε με τη σειρά Κύριος Μπέντλιν, ευχαριστούμε για τις παρατηρήσεις σας. Θα πρέπει να δούμε ότι ξεκάθαρα πρόκειται από όσα είπε η Επιτροπή και ο κύριος Σιόφνερ ότι το αποτέλεσμα της πρότασης δεν είναι σαφές. Αυτό τόνισα και εγώ στην εισηγησή μου ότι δεν γνωρίζουμε κατά πόσον αποσκοπεί πρώτα στο να έχει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα ή ου. Και αν, ναι, όπως είπε ο καθηγητής ε, Χέπνερ, τότε είναι σαφές ότι θα υπάρξουν περιπλοκές, προβλήματα όσον αφορά την ελευθερία του λόγου. Για σκεφτείτε τι θα γίνει όλοι αυτοί οι αγαπημένοι σας εκπρόσωποι του κυβισμού, πώς, τι, θα, τι θα είχε απογίνει για να χρησιμοποιούνται και να επαναχρησιμοποιούνται αυτά τα αποσπάσματα των ειδήσεων. Πώς όλα αυτά θα ρυθμιστούν με τις τρέχουσες εξαιρέσεις. Θα είναι μεγάλο πλήγμα για την ελευθερία έκφραση αν δεν επιτραπεί η χρήση από τον κόσμο αυτών των ε, αποσπασμάτων. Κύριε Κρέτσμερ, εκτός από το να απαντήσουμε, θα πρέπει να σχολιάσουμε αυτό που είπε ο καθηγητής Χέπνερ στην αρχή, ότι υπάρχει μια αντιστοιχία μεταξύ επιστημονικής έρευνας και εξυπηρετώντας ανάγκες κάποιου πελάτη. Είναι κάπως προβλητικό αυτό. Ε, τώρα είχαμε ως πελάτη έναν διαγωνισμό, ε, την, την πρόσκληση, οπότε μας είπε το Ευρωκοινοβούλιο και εμείς ε, ακολουθήσαμε με δημοσιεύσεις ε, με την μελέτη που φυσικά επιδέχεται ε, αναπαραγωγή. Μα αν είναι έτσι τα πράγματα και αν έτσι φέρει το κοινοβούλιο ως πελάτης, τι να κάνουν εδώ, τι, ποιος είναι ο ρόλος εδώ των επιστημόνων. βάση της μελέτης και αφετηρία ήταν ότι θέλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσουμε την πολυφωνία του τύπου. Και επίσης ως αφετηρία και αποδο... Ε, δεχτήκαμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν πλατφόρμες που να ωφελούν τους επαγγελματίες των ΜΜΕ. Έτσι είναι η προσέγγιση. Όμως είπαμε ότι δεν λειτουργεί το σύστημα τελικά. Όσο και αν έχουμε μικρό δείγμα, όμως είναι δείγμα ποιοτικό, γιατί αφορά κάποιους που κάθε μέρα παλεύουν σε αυτό το μέτωπο. Οπότε αφού μας είπαν ότι υπάρχει αποτέλεσμα, υπάρχει επίδραση στην ελευθερία της ε, έκφρασης, στην καινοτομία, στο πώς μπορεί να μπει στην αγορά, ε, δεν μπορούμε να λέμε τα ίδια και να μην υπάρχει κανένα αποτέλεσμα. Οπότε, αυτό είπαμε για τη μελέτη. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με αυτούς που κάνουν τις καινοτομίε, αυτοί οι οποίοι δουλεύουν και θέλουν μια τέτοια πολυφωνία στον τύπο και κάθε μέρα δουλεύουν εκεί. Να μιλήσουμε σε αυτούς και όπως ε, σας είπαμε από την, ε, τον όμιλο Spring για όλο αυτό το εισόδημα από τις δουλειές τους, τις ψηφιακές. Και αυτό κάθε χρόνο αυξάνεται, άρα καλά τα πάνε. Άρα σε εμά προσβλέπουν. Ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι έχουν γίνει πολλές ε, ακροάσεις και εργαστήρια όπου ακούστηκαν οι απόψεις αυτών που αναφέρεται. Ο κ. Χόπνερ έχει το λόγο. Ωραία. Θα ήθελα καταρχάς να αναφερθώ στην ελευθεροτυπία. Νομίζω ότι εδώ το copyright βοηθά, διότι αυτό που προστατεύεται είναι η συντακτική ευθύνη. Και η συντακτική ευθύνη είναι ακριβώς αυτό που οριοθετεί τις πραγματικές από τις ψευδείς ειδήσει. Επίσης, να αναφερθώ σε αυτό που είπε η κυρία Ρέντα. Φυσικά, ως ε, εκπρόσωπος του Safe Link, ε, της εκστρατείας Safe Link ε, δεν περιμέναμε τίποτα άλλο από το να διαστρεβλώσει τα πράγματα. εγώ πρέπει να σας πω ότι είπα ότι η, επίπτωση είναι ελάχιστη ε, στην, στους υπερσυνδέσμους. Το 2 με 3% δεν είναι σοβαρή επίπτωση όπως είπατε εσείς ότι υπάρχει. Επίσης Παραβλέψατε ε, τη σχέση ανάμεσα σε hyperlink και κείμενο. Κάτι που είναι ε, πλήρως, ε, διαστρέβλωση της ε, πραγματικότητας. Βεβαίως οι ανησυχίες που εκφράσατε ενδεχομένως ε, βασίζονται και σε κάποια ε, πραγματικά στοιχεία. Αλλά εγώ θεωρώ ότι το να πει κανεί ότι τα hyperlinks ε, αποτελούν κίνδυνο ε, είναι απλά κινδυνολογία. Άμα δείτε λοιπόν τον κύκλο εργασιών του ομίλου Springer και από πού προέρχεται στο ψηφιακό κόσμο, δεν είναι ειδήσει. Προέρχονται τα έσοδα από ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Ε, συγκριτικά πόρταλ για αγορές, πόρταλ έβρεση εργασία, αλλά όχι από τα ειδησογραφικά πόρταλ. Τα ειδησογραφικά πόρταλ δεν φέρνουν λεφτά, διότι το διαφημιστικό μοντέλο, το επιγραμμικό, δεν φέρνει χρήματα. Άρα η σύγκριση αυτή δεν είναι αιτιολογημένη. Αντίθετα, δείχνει ότι ο Άξελ Σπρίγκερ είναι απλώς στην ε, πρώτη γραμμή της ψηφιοποίησης Άρα δεν είναι ένα επιχείρημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον του. Όσον αφορά την ανεξαρτησία, εγώ δεν αμφισβήτησα την, την ανεξαρτησία σας, απλά αμφισβήτησα το αν, θα ήταν, αν είναι σωστό να ε, καλέσει κανείς να αξιολογήσει έναν επικριτή την ίδια την κριτική που ασκείται. Ο κύριος Καρόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να αφιερώσω τα δύο λεπτά που μου δίνετε για να επανέλθω στην έννοια του τεκμηρίου αντιπροσώπευσης ε, στο δικαίωμα δημιουργού και στα hyperlinks. Αυτό το τεκμήριο στο οποίο αναφερόμαστε σε μία από τις επιλογές της πρώτας της Εστονικής Προεδρίας βρίσκεται επίσης και σε ένα σχέδιο έκθεσης μου θυμίζει μια φράση του πρίγκιπα Σάλινα στο τέλος ε, ε, τη ταινία ε, η αναχώρηση πρέπει να αλλάξουν όλα ώστε να μην αλλάξει τίποτα. Στο τέλο δηλαδή θα τα αλλάξουμε όλα και στο τέλο δεν θα έχει αλλάξει τίποτα. Να σα εξηγήσω. Δηλαδή είτε οι εκδότε θα έχουν αγοράσει το δικαίωμα από τον δημιουργό και δεν χρειάζονται κανένα τεκμήριο εκπροσώπευση ή αντιπροσώπευση ή δεν έχουν αγοράσει το δικαίωμα από του δημιουργού, από του δημοσιογράφου. Σε αυτή την περίπτωση μία αγορά πώ μπορούμε να παραδεχτούμε ότι υπάρχει αντιπροσώπευση ενώπιον της δικαιοσύνης ενώ ο εκδότης ο οποίος θα εκπροσωπήσει αυτούς τους δημοσιογράφους ε, ε, ενώπιον της δικαιοσύνης σε ένα δικαίωμα το οποίο δεν κατέχει. Δεν υπάρχει ε, εκπροσώπηση στη δικαιοσύνη με τέτοιο τρόπο. Ποιος συμβαλόμενος θα συνάψει σύμβαση με μια επιχείρηση τύπου που το μόνο που του προσφέρει είναι μια εντολή αντιπροσωπευση για ένα δικαίωμα δημιουργού το οποίο δεν ξέρουμε αν υπάρχει τελικά μια εντολή που μπορεί εύκολα να ε, αποτελέσει το αντικείμενο ένσταση σε δικαστήριο. Βλέπετε πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η πρόταση λοιπόν και περί τι. Κάτι άλλο για τα hyperlinks τώρα. Κατά την άποψή μου είναι σημαντικό η νομοθεσία που θα υιοθετήσετε, αν την υιοθετήσετε, να μην εμποδίζει τη χρήση hyperlinks. Είναι πολύ σημαντικό να το προστατεύσετε αυτό. Αντιθέτως, όταν έχετε ε, φορείς που ονομάζονται crawlers, οι οποίοι ε, θα ταξινομήσουν, θα αναλύσουν και θα αξιοποιήσουν για έναν πελάτη που τους πληρώνει ε, hyperlinks, είναι φυσιολογικό οι άνθρωποι αυτοί να κερδίσουν χρήματα χάρη σε περιεχόμενο που έχουν φτιάξει με τεράστιες επενδύσεις από τις οι επενδύσεις, η, ε, εκδοτική οίκη. Το δικαίωμα αυτό της διανοητικής ιδιοκτησίας δεν συνίσταται πάντα στο επιτρέπω ή απαγορεύω, είναι και ένα δικαίωμα αποζημίωσης. Σημαίνει ότι ο εκδοτικός οίκος δεν θα απαγορεύσει ε, σε αυτή την περίπτωση τα hyperlinks, αλλά θα μπορεί να λάβει μια αποζημίωση. Αυτό είναι ένα κανόνα ο οποίο θα μπορούσε να αφορά ολόκληρο το κομμάτι τη διανοητική ιδιοκτησία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και εμεί. Να ευχαριστήσω όλου του διακεκριμένου ομιλητέ μα που βρέθηκαν εδώ μαζί μας σήμερα. Ευχαριστούμε που ε, μας προσφέρατε όλες αυτές τις πολύτιμες πληροφορίες. Η Επιτροπή συνεχίζει και κλεισμένο των θυρών. Να ζητήσω λοιπόν από όσους όλοι δεν έχουν το δικαίωμα να βρίσκονται σε μια συνεδρία και κλεισμένο των, των θυρών να αναχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν.